Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεδρία στην τονομία της Επιτροπής πριν από τις 10.30 όπου θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Θα πρέπει να εξετάσουμε δύο σημεία. Το πρώτο φορά, την τροποποίηση του άρθρου 90 του κανονισμού όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες. Θα θυμόσαστε ότι αυτό το αίτημα της εκθέσεως απευθύνθη στον πρόεδρο της Επιτροπής για το Διεθνές Εμπόριο διότι θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε ε, συμμόρφωση στον φάση διαδικασία στο Συμβούλιο. Σύμφωνα τον κανονισμό ζητήσαμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας και είπε ότι ο κανονισμός μας πρέπει να τροποποιηθεί, είπε τα αντίθετη νομική υπηρεσία, για να συμμορφωθεί με τις συνθήκες. Και τον συνάδελφο Μάρτιν ε, διορίσαμε ω εισηγητή, τον οποίο δίνω τώρα το λόγο. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της ΙΝΤΑ αλλά και ο κύριος Μπροκ, Πρόεδρος της ΑΦΕΤ. Επίσης ζήτησε έκθεση για το θέμα αυτό για λίγο διαφορετικούς λόγους. Θα επανέλθω. Προτείνω τρεις ε, τροποποίησεις του κανόνα 94, εδάφια 4, 5 και 6 λοιπόν. Και ο λόγος είναι οι κανόνες του Κοινοβουλίου να συμβαδίζουν με τη συνθήκη. Η τροπολογία 1 για το 1994. Οι κανόνες μας λένε ότι μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε μόνο όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα όταν έχουν καταλήξει συμφωνίες. Ο κύριος Μπροκ θεώρησε ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να πούμε κάτι και μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει εκπεφρασμένο δικαίωμα να εκφραστεί επί των διεθνών συμφωνιών. Ενώ βεβαίως ε, σύμφωνα με την πρακτική ε, δίνουν ε, γνώμη οι Επιτροπές, δεν το προβλέπουν οι κανόνες, οπότε θέλουμε να τροποποιηθεί για να συμβαδίζει με την πρακτική. Νόμιζα πως δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ίντα, που είναι από τη δική μου πολιτική ομάδα, τον κύριο Μορέιρα, που είπε ότι το τμήμα για την ε, γνωμοδότηση το δέχεται μεν, αλλά το να δίνει τη γνωμοδότηση μετά το τέλο των πραγματεύσεων και πριν καταλήξει η συμφωνία δεν είναι σοφρόν γιατί κατά τη γνώμη του, εφόσον η Επιτροπή έχει μονογράψει μια διεθνή συμφωνία, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Γιατί αφορά βεβαίω και του εταίρου. Αλλά θα μπορούσαμε εμεί ε, τότε να κάνουμε ε, σχόλια που δεν μπορούν να εφαρμοστούν και μετά στη διαδικασία σύμφωνης γνώμης ε, μπορεί να χρειαστεί να συμφωνήσουμε ενώ έχουμε εκφράσει πολλές επιφυλάξεις για την συμφωνία. Δεν θεωρεί λοιπόν ότι είναι σκόπιμη μια τέτοια γνωμοδότηση εφόσον έχουν λήξει οι διαπραγματεύσει και μονογραφηθεί συμφωνία μέχρι την τελική συμφωνία, τελική υπογραφή και δεν μπορούμε να αλλάξουμε πλέον τίποτα. Πρέπει να το συζητήσουν οι δύο πρόεδροι και θα με ενδιαφέρει και η γνώμη των συναδέλφων για τον κανόνα 95 τώρα για το κανόνα 90 παράγραφος 5 ναι μεν φαίνεται σαν μείωση των ε, αρμοδιοτήτων μας αλλά θα ε, ε, εναρμονίσει το κείμενο με τη συνθήκη δεν έχει λοιπόν ένα μήνυμα στην αρμοσμένη με τη συνθήκη τώρα για την παράγραφο 6 και εδώ θέλουμε να εναρμονίσουμε με την συνθήκη. Διότι τώρα όταν πρέπει να δώσουμε σύμφωνη γνώμη, οι κανόνε λένε ότι μπορούμε να απευθυνθούμε στο δικαστήριο για διευκρίνηση. Όταν γνωμοδοτούμε μόνο για μια διεθνή συμφωνία, οι κανόνε μα δεν μα επιτρέπουν να απευθυνθούμε στο δικαστήριο, αλλά η συνθήκη το επιτρέπει. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τι αρμοδιότητε μα ούτως ώστε οι κανόνε μα να μην μειώνουν αυτέ μα τι αρμοδιότητε. Τρει κανόνε, λοιπόν μετά την γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Τα, οι παράγραφοι 5 και 6 δεν δημιουργούν πρόβλημα. Έχουν επισήμω δικαίωμα να γνωμοδοτούν οι επιτροπέ. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα. Η μόνη συζήτηση είναι αυτή η συζήτηση για το τι θα μπορούμε να κάνουμε μεταξύ ε, λήξης των διαπραγματεύσεων και υπογραφή, Εάν θα μπορούσε κατά αυτή την περίοδο να σχολιάσει ή όχι το Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Υπάρχει κάποιο που θέλει να πάρει το λόγο όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Ορίστε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Μάρτιν. Η αιτιολογική έκθεση είναι αρκετά διεξοδική και είναι ευνόητες και οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Και πραγματικά είστε πολύ θαραλέος ε, που προωθείτε αυτή την έκθεση ενώ πλησιάζουμε στο τέλος της κοινοβουλευτικής μας και ο χρόνος μας πιέζει. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετές μεταφράσεις της έκθεσής σας σε όλες τις γλώσσες. Σε γλώσσες. Έχουμε μόνο 4-5 ε, γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά. Εν πάση περιπτώσει, παρά τη δυσκολία, θα κάνω μερικά σύντομα σχόλια. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό θέμα που θα πρέπει να θέσουμε για να βελτιώσουμε το άρθρο 90 των διαδικαστικών κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ποιο είναι το θέμα των γνωμοδοτήσεων ή της διαδικασίας έγκρισης η ε, σύμφωνης η σύμφωνη γνωμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι για το σχέδιο της ε, Διεθνούς Συμφωνίας ή δίνουμε την έγκρισή μας στην απόφαση του Συμβουλίου. Εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Ποιο είναι το αντικείμενο της δικής μας γνώμης. Στη διαδικασία υιοθέτηση ε, διεθνών συμφωνιών υπάρχουν αρκετά περίπλοκες διαδικασίες και εμείς θα πρέπει να δούμε σε ποια φάση δίνουμε την έγκρισή μας. Κανονικά θα πρέπει να δίνουμε για τη σύναψη της συμφωνίας. Βέβαια η διαδικασία έχει τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι εκεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το κείμενο της συμφωνίας. Αλλά αυτό το κείμενο θα πρέπει να το εγκρίνει το Συμβούλιο. Δηλαδή το, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο δύο προτάσεις. Μία για υπογραφή και μία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, για τη σύναψη της συμφωνίας. Η δεύτερη φάση ξεκινάει με την έγκριση από το Συμβούλιο της απόφασης ή του κανονισμού και με την υπογραφή της συμφωνίας. Και στην τελευταία φάση το Συμβούλιο υιοθετεί την απόφαση που ολοκληρώνει και συνάπτει τη συμφωνία. Εμείς έχουμε, έρχομαστε εδώ να παίξουμε έναν ρόλο μετά τη δεύτερη φάση, μετά τη δεύτερη απόφαση του, Συμβουλίου, εκεί που συνάπτει τη συμφωνία. Η απόφαση όμως αυτή για τη σύναψη της συμφωνίας θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο ή τη διαδικασία τη έγκριση τη σύμφωνη γνώμη. Γι' αυτό το άρθρο 95 θα μπορούσε να τροποποιηθεί. Θα πρότεινα όμω η τροπολογία να τροποποιήσει το draft agreement και να το αντικαταστήσει με το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας. Από το σχέδιο συμφωνίας να πούμε το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε ε, περιττές επαναλήψεις ε, υφισταμένων κανόνων. Να αποφύγουμε τις επαναλήψεις, γιατί επαναλήψεις για παράδειγμα έχει η τροπολογία που αφορά το 94 και ιδιαίτερα η τελευταία, παράγραφος, η τελευταία φράση που λέει κανόνε 49, 50 κτλ. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τέτοιε επαναλήψεις. Επίση, θα ήθελα κύριε Μάρτιν, αν γίνεται, να μου αναπτύξετε την ιδέα σα για την τροπολογία 2. Γιατί όταν υποβάλλεται αίτημα του, Ευρω... του Συμβουλίου προς το Κοινοβούλιο πηγαίνει στον Πρόεδρο και αυτό το παραπέμπει στην αρμόδια επιτροπή. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να το πούμε και πάλι αυτό στο άρθρο στον κανόνα 90. Υπάρχουν κάποια κρυφά προβλήματα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τις διεθνείς συμφωνίες. Και αν ναι, ποια είναι. Γιατί επισημαίνουμε κάτι τέτοιο στην τροπολογία 2. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι ε, φαντάζομαι ότι η προσωρινή συμφωνία ε, ή, ή μια διαδικασία μπορεί να είναι περίπλοκη, αλλά θα πρέπει θα πρέπει να διαρωτηθούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε όντως μία έκθεση για το θέμα αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να επαναλάβετε την πρότασή σας για το 94 ή το 95, 90 παράγραφος 5. Τι διατύπωση προτείνετε για το 95. Είπατε ότι θέλετε να διορθώσουμε τη διατύπωση του 90 παράγραφος 5. Εσείς προτείνετε να αντικαταστήσουμε τον όρο agreement, συμφωνία. Ή μάλλον εγώ προτείνω να αντικαταστήσουμε τον όρο σχέδιο συμφωνίας που προτείνει το αρχικό κείμενο από το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη συμφωνίας. Έχει νόημα αυτό που λέω. γιατί το σχέδιο συμφωνίας είναι πιο γενικό. Καλύτερα να πούμε σχέδιο απόφασης για τη σύναψη συμφωνίας. Είναι πιο ειδικό και αναφερόμαστε, εξειδικεύουμε τη φάση της διαδικασίας που μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό, ο κύριος Νταφ, για το σημείο αυτό. Εάν τροποποιήσει κανείς το 95, δεν είναι σχέδιο απόφασης, είναι η απόφαση για το σχέδιο συμφωνίας. Δεν είναι σχέδιο απόφασης. Για το βασικό θέμα, αν ο κύριος Μπροκ ή ο κύριος Μορέρα έχουν δίκιο από τις αντίστοιχες επιτροπές τους, αυτό συνεπάγεται ότι η φύση εμπορικής συμφωνίας διαφέρει από μια πολιτική συνθήκη συμφωνία. Από την οπτική γωνία της ΑΦΕΤ είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να μπορεί να εκφράζεται επί των διαφόρων λεπτομεριών και των αποχρώσεων μιας ε, διεθνούς ε, συμφωνίας. Άλλος που να μιλήσει, δεν υπάρχει άλλος. Α, θέλει να πει κάτι ο συνάδελφος Μάρτιν ακόμα, αν θέλει να δώσει απαντήσεις. Για το τελευταίο θέμα του κυρίου Νταφ, πρέπει να πω ότι θέλω να ε, αναφέρω όλες τις απόψεις ε, που υπάρχουν. Στην έκθεση Άκτα, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε το κείμενο, αλλά μια σαφής άποψη του Κοινοβουλίου μετά την ε, μονογραφή θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή να διευκρινίσει την κατάσταση και θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετική κατάληξη του θέματος αυτού. Άρα έχει κάποια ουσία ε, να μπορούμε να εκφραστούμε ακόμη και μετά τη μονογραφή. Για την παράγραφο 5 τώρα. Και αυτό που είπε ο κ. Γιούτσες. Ο λόγος για τη διατύπωση είναι για να ξεπεράσω το πρόβλημα. Καλή το Συμβούλιο, ε, ε, συγγνώμη, αιτήματα από το Συμβούλιο για τη γνώμη ή τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, άρα δεν εξετάζουμε τι είδος γνωμοδότηση. Εφόσον μας ζητήσει επισήμως το Συμβούλιο, να τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Δεν τροποποιούμε την υπάρχουσα διαδικασία. Αλλά μπορούμε να το ξαναδούμε αν επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Καλώς. Αυτή η έκθεση θα πρέπει να εγκριθεί, να ψηφιστεί στις 18 Μαρτίου στη συνεδρίαση. Μπορούμε να καθορίσουμε το χρόνο για τις τροπολογίες πολύ κοντά, 20 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις λοιπόν, αυτή είναι η απόφασή μας. Καλώς, ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Πάμε στην έκθεση του συναδέλφου Γκουαλτιέρη όσον αφορά την διοργανική συμφωνία που αφορά το Μητρό της Διαφάνειας. Η ομάδα εργασία δημιουργήθηκε από το Προεδρείο. Συμμετείχαν πέρα από τον υποφαινόμενο ο κύριος Γκουαλτιέρη και ο κύριος Ταρκόσκι. Αυτή η συμφωνία, αυτές οι διαπραγματεύσει, μάλλον ολοκληρώθηκαν με μια έγκριση το αποτελέσμα της πλευράς του Προεδρείου του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 127 η Επιτροπή μας θα πρέπει να, να το υποβάλει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Ο κ. Γκουαλτιέρη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Με αυτή την έκθεση πρέπει να πω ότι είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που οδήγησε σε τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά το Μητρό Διαφάνειας και αυτό υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο το κείμενο και ο στόχος της εκθέσεως πάνω απ' όλα είναι να αντικατοπτριστεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων όπου συμμετείχε και ο ίδιος ο εισηγητής και θέλαμε και από την άλλη να μην περιορίσουμε με συμβολογραφικό τρόπο αν θέλετε να αναπαράγουμε μια διοργανική συμφωνία με αυτόν τον τρόπο και είχαμε σαν στόχο μάλιστα να συμπεριλάβουμε πτυχές δύο προσεγγίσεων. Πρώτα απ' όλα, διαδρομή προς ένα υποχρεωτικό μητρό, πορεία προς ένα υποχρεωτικό μητρό και δεύτερο σενάριο, δεύτερη προσέγγιση που εμπεριέχει έκθεση όσον αφορά διάφορες στοιχές ερμηνευτικές όσον αφορά κάποιες καινοτομίες της συμφωνίας. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, Το Κοινοβούλιο κατ' παρελθόν τοποθετήθηκε υπέρ ενός υποχρεωτικού μητρώου. Αυτή η έκθεση εκ νέου προτείνει την ίδια προσέγγιση, ακόμα πιο περιοριστικά θα έλεγα, καθορίζοντας όχι μόνο ενδεχόμενες δυνατές διαδικασίες, αλλά και προθεσμία, deadline, που συζητήθηκε εξάλλου και με την ίδια την Επιτροπή τότε στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ανανέωση της συμφωνίας. Όπως σημειώνεται, όσον αφορά το θέμα αυτό, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αρχών και των εξουσιών που αναφέρει συνθήκες, διότι το άρθρο 11, παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ένωση, κατά την άποψή μου, σαφώς καθορίζει το στόχο που έχει ο διάλογος, ο διοργανικός, ο διάλογος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με την κοινωνία των πολιτών και με τις ενώσεις που τους εκπροσωπούν. Πρέπει να είναι όχι μόνο τακτικός και ανοιχτός αυτός ο διάλογος, αλλά και διαφανής. Υπάρχει σαφής αναφορά ενός στόχου. Οι στόχοι θα πρέπει να συνοδεύονται και από σαφή ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Από αυτή την έποψη οι συνθήκες οι παρούσες δεν θα επέτρεπαν μια εισαγωγή, μια θέσπιση ενός υποχρεωτικού μητρώου, αν και το άρθρο 352, η ρήτρα ευελιξίας όπως αποκαλείται, επιτρέπει την ανάθεση στην Ένωση Εξουσιών για την επίτευξη στόχων που καθορίζουν ήδη συνθήκες. Γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2016 να υποβάλει μια πρόταση βάσει του άρθρου 352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού μητρώου ή εναλλακτικά ε, εάν υπάρξει διαδικασία μεταρρύθμισης των συνθήκων να συμπεριληφθεί εντός συνθήκης η δημιουργία μιας ad hoc νομικής βάσεως για να θεσπίζεται ένα υποχρεωτικό μητρό. Είναι μια ισχυρή ένδειξη θα έλεγα, είναι μια από τις δύο ε, συνεισφορές που προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στη συμφωνία, μέσω της συμφωνίας η δεύτερη προσέγγιση αφορούσε την ερμηνεία, όπως σας είπα, των καινοτομιών που εισάγονται συμφωνία. Ε, θα πρέπει ακροθυγώς να αναφέρω κάποια σημεία. Διενεμήθη συμφωνία. Όλοι μπορείτε να σημειώσετε τις βελτιώσεις που στα πλαίσια του εθελοντικού μητρώου που βασίζεται περισσότερο σε κίνητρα παρά σε δεσμεύσεις Θέτει όμως παρόλα αυτά, ακόμα και εκεί τίθενται κάποια όρια, παρόλα αυτά επιφέρονται σημαντικές βελτιώσεις μέσω της συμφωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο Βίλαν που διεξήγαγε πάρα πολύ καλά τις εργασίες, διοργάνωσε πάρα πολύ καλά τις ε, εργασίες της πραγματευτικής ομάδας. Και ευχαριστώ βέβαια και όλους τους ε, άλλους συναδέλφους της ομάδας εργασίας. Και ευχαριστώ και τη γραμματεία. Η νέα συμφωνία πάνω απ' όλα εισάγει μία ενίσχυση και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Μητρώου, διευκρινίζοντας ότι πρέπει μέσω θα πρέπει να καταχωρούνται μέσω των κινήτρων ανεξάρτητα από εκεί που διεξάγονται οι δραστηριότητε των ομάδων πίεση, γίνεται καταχώρηση και αναφέρεται και το έμεσο lobbying που συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου. Και υπάρχει και άλλη ισχυροποίηση, δηλαδή ότι η καταχώρηση θα πρέπει να συνδέεται με τις δραστηριότητε που έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλά και αυτές που προετοιμάζονται. Και τέλος, υπάρχει και μια ενίσχυση, μια διευκρίνηση μάλλον που αφορά τα όρια ε, εξαίρεσης ε, του, του επαγγέλματος του νομικού που αυτή η εξαίρεση συνδέεται με τον τύπο δραστηριοτήτων που διεξάγει ένας ε, νομικός, όχι από το ίδιο του το καθεστώς, τη θέση του, αν ασκεί μια δραστηριότητα στα πλαίσια του ρόλου ενός δικηγόρου είναι άλλο. Αν είναι νομικός, αλλά δίνει συμβουλές, υποστηρίζει τις δραστηριότητε λόμπινγκ, εμπίπτει στο μητρό. Αυτό έχει και συνέπειες στις οποίες θα αναφερθώ σύντομα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εφαρμογή της συγκεκριμένης διευκρίνησης. Ενισχύουμε και την αναφορά τα κίνητρα. Η νέα συμφωνία λέει ότι τα κίνητρα δεν αποτελούν δυνατότητα. Πρέπει να εισαχθούν και να ενισχυθούν αυτά τα κίνητρα. Διότι τα κίνητρα σε ένα μη υποχρεωτικό σύστημα είναι, είναι ο κορμός, είναι η καρδιά. Οπότε τα κίνητρα είναι αποφασιστική σημασίας για την εύρυθμη ε, λειτουργία ενός μητρώου ε, διαφάνειας μετά τονίζουμε και υπογραμμίζουμε τα μέτρα της διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση μη σεβασμού των συμφωνιών και τέλος το παράδειγμα 2 θέλω να αναφερθώ ότι αναφέρεται η διαδικασία για τη χορήγηση πληροφοριών όλοι οι πελάτες που συνδέονται με τεστεριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ε, του πλαισίου αυτού πρέπει να αναφέρονται. Αυτές είναι οι καινοτομίες της συμφωνίας. Βεβαίως δεν είναι τέλεια συμφωνία, είναι καρπός διαπραγματεύσεων μεταξύ διαφορετικών φορέων και προφανώς δεν είναι υποχρεωτικό το Μητρό, μόσα συνεπάγεται αυτό, όμως αποτελεί ένα βήμα προόδου, μια βελτίωση. Στο ψήφισμα που επισυνάπτεται στη συμφωνία θέλουμε να δώσουμε κάποιες περαιτέρω ερμηνευτικές διευκρινήσεις πάνω απ' όλα στο τελευταίο σημείο που συνδέεται με το παράτομα 2 ε, θα πρέπει να αναφέρεται υποχρέωση για τα υποκείμενα που καταγράφονται, που καταχωρούνται να αναφέρουν όλους τους πελάτες τους και να διασυνδέεται ο κάθε πελάτης με την ασκούμενη δραστηριότητα. Αυτό είναι σημαντικό σημείο που αποτελεί μια τροποποίηση και ενίσχυση του κειμένου όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώρηση. Προσπαθεί η έκθεση μετά να ε, συμβάλλει στον ορισμό των μη ενδεδειγμένων συμπεριφορών, των απλεπών συμπεριφορών και σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να φέρουμε όλες τις τυπολογίες της παρέμβασης στην ιδιωτική ζωή, στην ιδιωτική σφαίρα, ακόμα και τις πιο μικρές παρεμβάσεις, έλλειψη επικοινωνίας όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων των εκπροσωπουμένων ε, πελατών και μετά όσον αφορά τους νομικούς εκτιμούμε την, το σαφέστερο ορισμό της συμφωνίας σε αυτό το θέμα και καλούμε τους δικηγορικούς συλλόγους της Ευρώπης, πώς να το πω, να υποστηρίξουν την προσέγγιση σε αυτό το πλαίσιο μέσω θετικών παραδειγμάτων που παραθέτουμε όσον αφορά ε, τους δικηγορικούς συλλόγους των Βρυξελών και του Παρισίου. Δίνουμε και κάποιες πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες που θα αξιολογήσει το Προεδρείο πώς θα εφαρμόσει αυτά τα σημεία όσον αφορά το σύστημα των κινήτρων, κίνητρα που μπορούν να είναι περαιτέρω διευκολύνσεις, από την άλλη όμως θα μπορούσαν και θα έπρεπε ίσως να ερμηνευθούν και σαν αντικίνητρα για εκείνον που δεν καταχωρείται στο Μητρό. Εν αυτή τη ενία δίνονται κάποια παραδείγματα στην έκθεση πέρα που ζητείτε να ενθαρρυνθεί η παλήθευση της εγγραφής και εξακρίβωση αυτής, αλλά αναφέρονται και περιορισμοί σύμφωνα με τις γενικές αρχές της λειτουργίας του Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση στα μη καταχωρημένα υποκείμενα να δίνεται δυνατότητα συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου μόνο σε καταχωρημένα υποκείμενα, να καλούνται ως αγορητές, ως ομιλητές σε ακροάσεις στις επιτροπές που μόνο οι καταχωρημένοι ομιλητές θα μπορούν να, να μιλήσουν. Θα πρέπει εξολογείται η δυνατότητα λοιπόν να δίνεται μια χορηγία μόνο σε περίπτωση των καταχωρημένων ομιλητών. Αυτές είναι διευκρινήσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο κατά την άποψή μας η συμφωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη και η έκθεση συμπεριλαμβάνει και εδώ σταματώ και θα μπορέσω να δώσω αργότερα άλλες λεπτομέρειες και λεπτομέρειες θα τις δείτε διαβάζοντας τη συμφωνία Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να πω, θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας και θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Βίλαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτή την δραστηριότητα αναθεώρηση συμφωνία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Γκαλτιέρη για την έκθεση αυτή που είναι πληρέστατη. Ο κύριος Σέφλιν ζήτησε το λόγο. Yes, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Γουαλτιέρη για την έκθεσή του. Έχω μερικές απορίες. Η έκθεση είναι εμπεριστατωμένη. Στην παράγραφο 6. Τώρα, είναι σημαντικό να αποκαλύπτεται η ταυτότητα όλων των πελατών. Πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Και στην παράγραφο 7 το θέμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Πολύ σωστό αυτό πολύ σωστή μνήμα. Κάτι που καλύπτεται εν μέρη είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε το πρόβλημα της άσκησης πίεσης από οργανώσεις που έχουν σχέσεις ε, με τρίτες χώρες, που δεν είναι ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διπλωμάτες. Βέβαια αποκλείονται, αλλά δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις περιπτώσεις. Αν δεν κάνω λάθος, όταν πήγαμε στην Ουάσιγκτον, το είχαμε συζητήσει ότι έχουν κάποιου διπλωμάτε διαπιστευμένου, ίσω ή εγγεγραμμένους στο Μητρό. Ίσως κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί έχουμε υποστεί πιέσει από τέτοιου διπλωμάτε που δεν έχουν εγγραφεί αλλά είναι διαπιστευμένοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αποκλείουμε σελίδιν αυτή την κατηγορία. Τέλο, παράγραφο 12. Έχω την αίσθηση και δεδομένου και του παραρτήματος ότι δίνει κίνητρα σε όλους να βρουν κάποιον για να τον εγγράψουν. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά μήπως έτσι επιβαρύνουμε τη διαδικασία καταγραφής. Γιατί, αν διαβάζω καλά την πρόταση, ο καθένας που θέλει να οργανώσει μια δημόσια ακρόση θα πρέπει να τους καταγράφει όλους. Ακόμη και αν έχουμε τη συμμετοχή μια οργάνωση μία φορά τη πενταετία, αν θέλουν να συμμετέχουν σε μία δημόσια κρόση πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι. Δεν νομίζω ότι είναι στόχο ε, αυτή τη πρόταση μία τέτοια υπερβολική επιβάρηση. Ίσως παρά είμαστε αυστηροί εδώ. Και τώρα, πώ ε, θα γίνει αυτό το φιλτράρισμα, πώ θα ε, ληφθεί απόφαση για το ποιο επιτρέπεται να γραφεί και ποιο όχι εννοείται μια προσωρινή εγγραφή, δηλαδή βραχυπρόθεσμη και μια συνοπτική διαδικασία, fast track. Αν θέλουμε να προσκαλέσουμε μια συγκεκριμένη οργάνωση, σε μια συγκεκριμένη δημόσια κρόση, μια φορά ανά πέντε χρόνια, ας πούμε. Δεν είναι σκόπιμο να έχουμε μια πιο συνοπτική διαδικασία για τέτοιε περιπτώσει. γιατί κάτι τέτοιο απαγορεύεται με την τρέχουσα διατύπωση. Και τέλο, μια διευκρίνηση στην παράγραφο 16. Τι θα πει non-institutional watchdog, δεν είναι σαφές αυτό. Μη θεσμικός φορέας παρακολούθησης επιθαρχίας. Ευχαριστώ και Σέπλιν. Ο κύριος Βίλαντ έχει το λόγο τώρα. Ähm, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ο οποίος κατόρθωσε να αναφέρει και να ταξινομήσει τα βασικά σημεία που μας απασχόλησαν στην συζήτηση. Τον ευχαριστώ λοιπόν που κατάφερε παρά την πίεση χρόνου θέλουμε ε, να έχουμε ένα αποτέλεσμα για την επόμενη θητεία η ομάδα εργασία άρχισε τις εργασίες τη λίγο μετά τις διακοπέ είχε 10 συνεδριάσει και τα κατάφερε. Να πω τα εξή. Για τα σημεία 2 έως 5. Ο εισηγητής παρουσίασε πολύ σωστά τον προβληματισμό μας. Γιατί ξέρετε είναι σαν να έχουμε και να μην έχουμε νομική βάση. Το άρθρο 252 κατά γενική εκτίμηση δεν είναι το πιο κατάλληλο. Γιατί για πολύ καιρό δεν υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο και τα άλλα άρθρα δεν επαρκούν. Και αυτό πιστεύουμε ότι η Κομισιόν πρέπει να μας βοηθήσει να ασκήσουμε ε, λίγο περισσότερη ε, πίεση για να αλλάξουν κάπως οι συνθήκες, αν είναι δυνατόν. γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το Μητρό Διαφάνειας θα πρέπει να έχει μια καλύτερη νομική βάση. Και αυτό είναι το βασικό. Υπάρχουν διάφοροι που λένε ε, να είναι υποχρεωτικό αυτό το Μητρό, αλλά παραγνωρίζουμε έτσι ότι δεν μπορούμε απλά και μόνο να αποφασίσουμε ότι είναι υποχρεωτικό αυτό το Μητρό, γιατί αυτό έχει νομικές επιπτώσεις, συνέπειες. Και δεν έχουμε νομική βάση γι' αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποφασίσουμε ε, για πράγματα που έχουν ε, ευρείες νομικές επιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό που είπε αρχικά ο εισηγητής, ότι το άρθρο 11 παράγραφος 2 σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε πληροφόρηση, σε εκδηλώσεις που γίνονται στο Κοινοβούλιο. Εάν θέλουμε λοιπόν να είναι σαφές ότι θέλουμε να είναι υποχρεωτικό το Μητρό, τότε πρέπει να κάνουμε περισσότερα βήματα. Δηλαδή να πούμε ότι δεν υπάρχει νομική βάση και όσο πλησιάζουμε αυτό το αόρατο όριο, όπου δεν υπάρχει υποχρέωση αλλά και δικαίωμα για διάλογο, ε, δημιουργούμε πρόβλημα. Πρέπει να μείνουμε μακριά από αυτό το όριο. Για το 7. Πιστεύω ότι περιγράφεται πολύ καλά τι εννοούμε ανάρμοστη συμπεριφορά. Πιστεύω ότι στο μέλλον πρέπει να περιγράψουμε και άλλες καταστάσεις ή να τις ε, ορίσουμε καλύτερα. Πρόσφατα άκουσα ότι Μία συνάδελφος που ήταν εισηγήτρια διαμαρτυρήθηκε ότι έλαβε δεκάδες χιλιάδες email. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί κανείς να θεωρεί ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να πιέζουν έτσι τα μέλη του Κοινοβουλίου, ορισμένοι, που υποτίθεται ότι είναι συνομιλητές μας. Γιατί στην ουσία προσπαθούν ε, να σταματήσουν ε, τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, να πήξουν ε, τα σερβερ. Πρέπει λοιπόν να είναι η συμπεριφορά τους μετρημένη. Κάτι άλλο. περιγράφει ο εισηγητής στην, ε, στο, στην παράγραφο 10. Ξέρω ότι οι δικηγορικοί συλλογιστές και στο Παρίσι έχουν πει, έχουν πάρει αποφάσεις, ότι υπάρχουν τα κλασικά δικηγορικά γραφεία και τα μη κλασικά. Να το πω έτσι. Παίρνουμε δηλαδή ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο όπου κάθεται ένας δικηγόρος για να μπορεί να πει ότι να εδώ έχω το γραφείο μου και έχω όλα τα προνόμια του δικηγόρου. Αυτό είναι πρόσχημα. Από την άλλη, στην άλλη άκρη της κλίμακας υπάρχουν κράτη-μέλη όπου υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι περιορισμοί στο Σύνταγμα όπου δεν είναι δυνατόν, ακόμη και αν συμφωνεί ο πελάτης, ο δικηγόρος να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του πελάτου. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τόσο διαφορετικές ρυθμίσεις. Συζητώ λοιπόν με τους δικηγορικούς λόγους για να δούμε εάν θα ήταν δυνατόν να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει μια διαδικασία να μπορούμε υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας να δούμε εμείς γιατί δεν θα μπορούσε κάποιος δικηγόρος να γνωστοποιήσει την ε, ταυτότητα του πελάτου. Να κοιτάξουμε λοιπόν και να πούμε ναι, ναι, αιτιολογείται αυτή η εμπιστευτικότητα. Αλλά χωρίς ε, ε, νομική βάση δεν μπορούμε φυσικά να θίξουμε την εθνική νομοθεσία και πολύ λιγότερο τα εθνικά συντάγματα. Πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε περαιτέρω. Χαίρομαι λοιπόν για τη διατύπωση του 10, γιατί αντιμετωπίζει το πρόβλημα, χωρίς όμως να ξυπνά προσδοκίες που προς στιγμή δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε και το 12. Το ανέφερε ο συνάδελφος Σόπφλιν ήδη, όπου καλείται να εξετάσει και άλλα θέματα το Προεδρείο. Τα χαιρετίζω, αλλά το 12α μου δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες. Ο κάθε συνεργάτης, ακόμη και κατώτερου βαθμού θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται Νομίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το λοιπό προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να του περιλάβουμε όλου. Οποιοδήποτε που είχε απασχοληθεί ή είχε αναλάβει κάποια καθήκοντα, ούτως ή άλλως έχουμε τώρα το καθεστώ των βοηθών που μα επιτρέπει να διευκρινίσουμε την κατάσταση. Χαιρετίζω επίση την πρόταση του συναδέλφου Σέφλιν για του διπλωμάτε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλη μια ιδεολογική σκέψη την επόμενη φορά που θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτή τη φάση είναι δύσκολο να ε, βάλουμε και άλλα θέματα. Θα απαντήσει βέβαια ο Σνάλφος Γκουαλτιέρη σε αυτά που λέει ο Σνάλφος Σέπφλιν, αλλά η, δυνατό, η ιδιότητα προσώπου να, να συμπεριλαμβάνει στην Επιτροπή λέει εκεί ότι οι ομιλητές ε, σε ακροάσεις. Πρόκειται για συμμετέχοντες λοιπόν δεν μπορούμε σε όσοι συμμετέχουν σε συζητήσει στρογγυλή τραπέζη να αφαιρούμε το δικαίωμα να σχολιάσουν. Να πρέπει και αυτοί να εγγραφούν είναι λίγο ωριακό. Όσο μίλησε και για τα οικονομικά θέματα, στο σημείο 17 συγκεκριμένα, αναφέρουμε ότι δεν έχουμε επαρκές προσωπικό και ότι η Κομισιόν δεν έχει τη βούληση να ε, αποσπάσει αρκετούς υπαλλήλους για αυτό το κοινό μητρό. Οπότε ο έλεγχος μπορεί να γίνεται μόνο πολύ περιορισμένα των στοιχείων που μας υποβάλλονται. Και γι' αυτό ακριβώς και δικαίως αναφέρουμε στο άρθρο 16 το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Αν κάποιος ε, απ' έξω διαπιστώσει κάτι θα πρέπει να μπορεί να μας ενημερώσει να μπορεί να κάνει την αναγκαία καταγγελία. Και μετά για την ε, διαχείριση αυτών των καταγγελιών ε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Χαιρετίζω λοιπόν την έκθεση αυτή όπως έχει υποβληθεί και με κάποιες ε, διαφοροποιήσεις, κάποιες αναδιατυπώσεις θα μπορούσα να τη δεχτώ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος διότι διευκρινίζει σαφώς ότι δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουμε κάτι χωρίς νομική βάση γιατί είμαστε φυσικά κοινότητα δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίλεντ. Πολλά ε, ήταν αποτελέσματα της ομάδας εργασίας. Ε, λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν τα όσα είπα τις παρατηρήσεις σας. Ο συνάδελφος ο κ. Χέφνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Γουαλτιέρη, τον εισηγητή, τον κύριο Βίλαν και όλους όσους συμμετείχαν για την εργασία που επιτελέστηκε στην ομάδα εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Είναι αναγκαίο να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι δεν εργαζόμεθα για μας τους ίδιους, αλλά για τους πολίτες. Δεν είμαστε οι πολίτες, είμαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών και οι πολίτες τους οποίους εκπροσωπούμε. Έχουν δικαίως, κατά τη γνώμη μου, δικαίωμα να απαιτούν η εργασία μας να είναι διαφανής, να μπορούν να την παρακολουθήσουν. Και ιδιαίτερα όταν λαμβάνουμε αποφάσεις που αφορούν ε, το καλό των πολιτών, να έχουμε ακριβώς το καλό των πολιτών ως κριτήριο και όχι τα συμφέροντα ομάδων πίεσης, ε, επιχειρήσεων κτλ. Όλα αυτά είναι αναγκαία αν θέλουμε η κοινή γνώμη να εκτιμά την εργασία μας γιατί στο παρελθόν υπήρξαν δυσάρεστες εξελίξεις, σκάνδαλα και η κοινή γνώμη θέλει να υπάρχει μέγιστη διαφάνεια. Το Μητρό Διαφάνειας, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχουν όλα τα κοινοβούλια τέτοια Μητρώα. Αλλά όπως είπαν και οι προηγούμενοι, υπάρχουν σημεία που είναι ανεπαρκή. Και το ζήτημα είναι ότι είναι τα χέρια μας δεμένα. Σε αυτούς που λένε λοιπόν, μα γιατί δεν αποφασίζετε ότι όλα αυτά είναι υποχρεωτικά, δεσμευτικά για όλες τις επαγγελματικές ομάδες και να λύσατε το πρόβλημά σας. Οι Γκουαλτιέρη και Βίλαντ σωστά τόνισαν ότι υπάρχουν ε, νομικά όρια τα οποία από μόνοι μας με αποφάσεις του Κοινοβουλίου μόνο και μόνο με διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Χρειάζεται αλλαγή των συνθήκων, μία άλλη νομική βάση στη συνθήκη. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα τον Ρομπέρτο Γκουαρτιέδη που στις παραγράφους 1 έως 4 κατέστησε σαφές ότι αυτή είναι, αυτό είναι το πρωταρχικό μας αίτημα. Θέλουμε αυτή, αυτό το μητρό να γίνει τόσο δεσμευτικό, τόσο υποχρεωτικό, όπως ακριβώς το επιθυμούμε, όπως ακριβώς το απαιτούμε. Αλλά είναι λοιπόν, όπως είπα, προς στιγμή δεμένα τα χέρια μας και γι' αυτό εργάστηκε η ομάδα εργασίας και κατέληξε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί αυτό το αποτέλεσμα είναι το, σε αυτή τη φάση, εφικτό. Ορισμένοι θεωρούν πολύ ότι είναι ανεπαρκές. Η δική μου άποψη είναι ότι εργαστήκαμε ε, μακροχρόνια και επίπονα και αυτό το οποίο αποφασίσαμε, αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι το εφικτό. Για να κάνουμε όσο δυνατόν πιο διαφανές, όσο δυνατόν πιο υποχρεωτικό το μητρό αυτό. Υποστηρίζουμε λοιπόν ανεπιφύλακτα το αποτέλεσμα αυτό. Θα περάσουμε και στις ψηφοφορίες δεν θα περάσω τώρα στις ε, λεπτομέρειες, ε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, το είπαν οι προηγούμενοι. Για ένα σημείο μόνο θέλω να συμπληρώσω κάτι. Ξέρετε βεβαίως ότι είμαι πρόεδρος ε, της Συμβουλευτικής Επιτροπής που ασχολείται με την τήρηση των κανόνων μας, των κανόνων που έχουμε θεσπίσει με τον κώδικα διοντολογίας και των οποίων πρέπει να απαιτήσουμε την τήρηση, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι τιμούν το αξιωμά τους. Και ότι το σώμα μας τηρεί θεμελιώδεις κανόνες. Με βάση λοιπόν αυτά θα πρότεινα στην παράγραφο 7 όπου μιλάμε για ανάρμοστη συμπεριφορά να ε, συμπεριλάβουμε τρεις σαφείς ορισμούς. Τι σημαίνει ανάρμοστη συμπεριφορά. Η πρότασή μου θα ήταν και θα κάνω και την αναγκαία τροπολογία, πρέπει να σκεφτώ τη διατύπωση. Η πρότασή μου θα ήταν λοιπόν να αναφερθούμε και σε οικονομικά ωφέλη που μπορεί να λαμβάνουν βουλευτές από ομάδες πιέση άτομα. Γιατί είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και νομίζω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τέτοια συμπεριφορά που θίγει την ε, ανεξαρτησία του βουλευτή ή τουλάχιστον ε, την θέτει υπό ισχυρή αμφιβολία από αυτούς ε, που χορηγούν οικονομικά ωφέλεια ή ωφέλη, συγγνώμη. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεωρείται ανάρμοστη συμπεριφορά. Θα πρέπει να ισχύει αυτό λοιπόν και για δώρα πάνω από ένα αρκετά ευτελές ποσό και για κάθε άλλου είδους ωφέλη. Αυτά λοιπόν. Επιφυλασσόμεθα να κάνουμε και άλλες τροπολογίες, αλλά καταρχήν συμφωνούμε με αυτό το αποτέλεσμα των συζητήσεων των πολιτικών ομάδων και στα πλαίσια αυτών που θεωρούμε ότι είναι εφικτά σε αυτή τη φάση και τονίζουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμεθα ως Κοινοβούλιο για ένα πραγματικά υποχρεωτικό μητρό και να κάνουμε και την έκκληση στην Κομισιόν μέσω πρώτα αλλαγή των συνθήκων να δημιουργήσει αναγκαίε προποθέσει. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Νταφ στην τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω τη συμφωνία αυτή γιατί θα πρέπει ήδη από το 2010 όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για το Μητρό Διαφάνειας ε, σε αυτό το αποτέλεσμα να είχαμε καταλήξει. Και νομίζω ότι πραγματικά διδαχθήκαμε από την εμπειρία της ε, χρήσης ε, και εφαρμογής αυτού του Μητρό τη τελευταία διετία, τριετία. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να προσβλέπει σε πολύ υψηλέ προδιαγραφές ε, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και μάλιστα να βελτιώσει και τις πρακτικές των εθνικών κοινοβουλίων που πολύ συχνά είναι αξιοθρύνητες ε, για θέματα τέτοια. Πάντως σίγουρα πιστεύω ότι μια και πλησιάζουμε σε μια αναθεώρηση των συνθήκων, καλό θα ήταν να εξετάσουμε το άρθρο 298 που μιλάει για ανοιχτό, α, η ανοιχτή αποτελεσματική και ανεξάρτητη ε, ευρωπαϊκή διοίκηση. Βέβαια δεν πιστεύω ότι μια τέτοια ορολογία αρκεί για να έχουμε μια πιο δημοκρατική ένωση και μια καλύτερη δημοκρατική παιδεία. ή ότι κάτι τέτοιο ισχύει τώρα περισσότερο από ότι κατά τη σύνταξη της σχετικής ρήτρας της συνθήκης. Πιστεύω ότι το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει τεράστια ευθύνη κατά την εφαρμογή του διοντολογικού κώδικα και θα έπρεπε το Προεδρείο να εφαρμόσει αυτό το διοντολογικό κώδικα πολύ πιο αυστηρά από ό,τι στο παρελθόν. Και θα ήθελα να επενέσω τον κύριο Βίλαντ για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει για την αυστηρότερη αυτή εφαρμογή του κώδικα διοντολογίας. Και επίσης Πιστεύω ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν και θεμητές και αθέμητες πρακτικές ε, νομικές ε, και δικηγορικές πρακτικές, το ίδιο ισχύει και για τη διπλωματία. Υπάρχουν και θεμητές και αθέμητες συμπεριφορές. Και πραγματικά λυπούμαστε για την ε, ρεβασιστική συμπεριφορά μερικές φορές ε, που ε, υιοθετούμε για κάποιες ε, εκθέσεις έργων τέχνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ε, μια πρόσφατη για το Αζερμπαϊτζάν, την οποία ήμουνα παρόν. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο σχολαστικοί και να απορρίπτουμε ε, μερικές, ε, μερικά πολιτικά διαβήματα που είναι καθαρά δημοσιοσχεσίτικα και τέτοιες συμπεριφορές δυστυχώς εφαρμόζουν ορισμένες τρίτες χώρες. Αυτά, αλλά γενικώ η ομάδα μου συμφωνεί με το ψήφισμα. Αν ο κύριος Γκαλτιέρη θέλει να πει δύο, δύο λόγια, αν ήδη απαντήσω, αν πιστεύει χρειάζεται, ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατος. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα όλους τους συναδέλφους για όσα είπαν. Τους ευχαριστώ που εξετίμησαν το επιτελεστέν έργον. Να δώσω κάποιες σύντομες απαντήσεις στο ερώτημα του κυρίου Σέφλινγκ. Οι ξένοι διπλωμάτες αποτελούν μεγάλο πρόβλημα το συζητήσαμε. Κάτι που δεν σχετίζεται άμεσα με τους διπλωμάτες, αλλά μικτούς φορείς θα μπορούσε να καλύπτεται από το τελευταίο τμήμα του παραρτήματος 1. Το θέμα των διπλωματών βεβαίως δεν καλύπτεται και θα πρέπει να το σκεφτούμε. Συμφωνώ είναι μεγάλο ζήτημα αυτό πρέπει να είναι σαφής η διάκριση μεταξύ ε, εξωτερικών σχέσεων, εξωτερικής πολιτικής και των δραστηριοτήτων των ομάδων πίεσης. Σίγουρα πρέπει να το αναλύσουμε περαιτέρω. για τις πολύ, τους πολύ αυστηρούς όρους για τη συνδιοργάνωση ακροάσεων Δεν λέω ότι όποιος οργανώνει ή συνδιοργανώνει μια εκδήλωση πρέπει να καταχωρείται, να εγγράφεται, αλλά αν καλύπτεται το πεδίο εφαρμογής συμφωνίας, η εκδήλωση, θα πρέπει κάτι τέτοιο να ισχύει. Βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολικής φόρτωσης του συστήματος, χρειάζεται σωστή ισορροπία. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλο άχθος. Καλύτερα να έχουμε περισσότερη διαφάνεια παρά το αντίθετο. για το Watchdog ήδη οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με τη διαφάνεια συμβάλλουν σημαντικά. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα ήταν ευπρόσδεκτος ο ρόλος τους και τους ενθαρρύνουμε να παίξουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Για να συνεργαστούν με το Μητρό χωρίς αυτό να αντιβαίνει στο αίτημά μας να ενισχυθεί και η δομή και το προσωπικό αυτής της κοινή γραμματείας Μητρώου Διαφανείας, το οποίο προσωπικό βεβαίως εργάζεται θαυμάσια και θέλω να τους ευχαριστήσω για την μέχρι τούδε συμβολή τους στην έκθεση. Αυτό που είπε ο κύριος Βίλαντ. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσω, συμφωνούμε. μερικές παρατηρήσεις για το θέμα της νομικής βάσης και το υποχρεωτικό μητρό. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό τμήμα της έκθεσης. Υπογραμμίζω και πάλι ότι συμφωνούσα με την προθεσμία της Κομισιόν. Υπάρχουν δύο επιλογές. Μία είναι να τροποποιηθεί η συνθήκη, ούτω ώστε να δημιουργηθεί συγκεκριμένη για αυτό το θέμα, νομική βάση, αλλά το 352 θα μπορούσε ήδη να επιτρέψει τη δημιουργία ενός δεσμευτικού μητρώου. Βέβαια το 352 είναι βαριά διαδικασία. Αλλά είναι διάταξη ε, της ισχύουσας συνθήκης. Αλλά πρέπει η Κομισιόν να κάνει πρόταση. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι εκτός εάν μέσω αλλαγής της συνθήκης για να δημιουργηθεί η ειδική νομική βάση που θα ήταν η βέλτιστη επιλογή, σε κάθε περίπτωση πριν το 2016 η Κομισιόν πρέπει να υποβάλει πρόταση, ούτω ώστε να υπάρξει αρμοδιότητα για δημιουργία με βάση του άρθρου 52 υποχρεωτικού Μητρώου Διαφάνειας. Αυτό ζητούμε ως Κοινοβούλιο, εάν εγκριθεί βεβαίως η έκθεση. Αυτό ζητούμε να κάνει η Επιτροπή. Α, να προσθέσω όμως επίσης ότι προσβλέπουμε σε περαιτέρω διευκρίνηση του ορισμού της ανάρμοστης συμπεριφοράς από τους πρασίνους. Αυτά που γράψαμε εδώ δεν είναι ο ορισμός της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και άλλα στοιχεία στον ορισμό λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έχουμε ήδη καθορίσει και συμφωνήσει. Οτιδήποτε βελτιώνει αυτές τις τρεις ε, ήδη ε, συμφωνημένες προτάσεις θα ήταν πολύ χρήσιμο και ευπρόσδεκτο. Τέλος, τέλος. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Τζέραλντ Βεβαίω, συμφωνώ με αυτό που είπε ο ε, είμαστε υποχρεωμένοι να εκπροσωπούμε του πολίτε με το πιο διαφανή τρόπο. Η βελτίωση λοιπόν ε, του Μητρώου Διαφάνεια και ένα οδικό χάρτη ε, προ ένα υποχρεωτικό τέτοιο Μητρό είναι σημαντικό τμήμα των υποχρεώσεών μα και του ρόλου μα ω εκπροσώπων των πολιτών τη Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε τι προθεσμίε να να εγκρίνουμε την έκθεση στις 18 Μαρτίου για τις τροπολογίες 20 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία. Συμφωνούμε, ούτως απεφασίστη. Πάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Έχουμε τρεις εκθέσεις να ψηφίσουμε. Η πιο μακροσκελής είναι η έκθεση Ρανζέλ όσον αφορά την εφαρμογή της συνθήκης της όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση Ρανζέλ, όσον αφορά τη συνθήκη της Αβώνα, όσον αφορά την εφαρμογή της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν διάφορες συμβαστικέ τροπολογίες. Ψηφίζουμε τη συμβαστική Α. Υπέρ. Δυνατάσεως της Κατά. Τέσσερις ψήφια εναντίον. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην τροπολογία 22. Όλες οι άλλες βλέπετε καλύπτονται από τη συμβαστική. Τροπολογία 22. Υπέρ παρακαλώ. Σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και η τροπολογία 22. Πάμε συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Τέσσερις εναντίον. Άποχες. Καμία. Εγκρίνεται η συμβαστική Β. Αυτό μας επιτρέπει να πάμε να ψηφίσουμε την τροπολογία 30, διότι όλες οι άλλες που προηγούνται καλύφθηκαν. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Fox Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 33 και 34 πρέπει να ψηφιστούν. Κάνουμε τον έλεγχο έτσι να είμαστε σίγουροι. Ψηφίζουμε την 33. Φόξ. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Νταφ. Υπέρ. Κατά. 11, κατά, οπότε δεν εγκρίνεται. Συμβιβαστική, σι λατινικό. Α, είχαμε μία αποχή, ζητώ συγγνώμη. Μία αποχή είχαμε πριν. Αποφασιστική τη αυτή η περίπτωση. Συμβιβαστική, σί λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 38. Αόκι Ζήλστρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έτσι μπορούμε να πάμε στην τροπολογία 43. ραντ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασ... Συγγνώμη, τροπολογία 44 και 45 μαζί είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική έψιλον ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην τροπολογία στη συμβαστική F λατινικό διότι επεσήρθη η τροπολογία 50 και άλλες εκαλύπτοντο. Συμβαστική F λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. καταπίπτουν οι άλλες. Πάμε στη συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και αμέσως μετά έχουμε τη συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε μπορούμε να πάμε. Έχει αποσυρθεί 55 και πάμε επειδή καλύπτονται οι άλλες, στην τροπολογία 62. 62 υπέρ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να μετρήσουμε. Απορρίπτεται. Συμβαστική γιώτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 68 ντάφ υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε. Γιούρι. Λοιπόν, υπέρ. Στην παράγραφο 1. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 2 που αφορά την παράγραφο 13α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλύπτεται λίμπε 1. Πάμε στη Γιούρι 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι 10, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 9, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 και 81 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε την 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 Σάερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική L λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 87 διότι άλλες καλύπτονται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 καλύπτεται η εννέα από τις άλλες 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 7 υπέρ. Κατά. Θα μετρήσουμε. εγκρίνεται. Η Τζούρι 7. Πρόεδρε, λέει ο Νταφ, πρέπει να ακολουθήσουμε την ηλεκτρονική μέθοδο που συνήθως ε, λειτουργεί. Μήπως μπορούμε να κάνουμε επαλήθευση όσον αφορά τη Τζούρι 7. Νομίζω ότι είναι σωστό να δεχτώ το έτοιμά σας. Ας γίνει λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε λοιπόν τη Λίμπε 12, λέει ο Πρόεδρος. Α, Τζούρι 7. Τζούρι 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκατέσσερις ψήφοι υπέρ, εννέα ψήφοι εναντίον, μία αποχή, άρα εγκρίνεται. Καλά τα είδα. Λίμπε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κατέπεσε η άλλη γιατί εγκρίθηκε 7. Πάμε στη τζούρι 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τζούρι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 Φόξιπερ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα τη Ίντα, 11 μόνο ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ίντα 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 8 κατέπεσε Πάμε λοιπόν στη συμβαστική N. Νίλατη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική μη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε ψηφίζουμε τώρα. Την τροπολογία 96. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 'Κατέπεσε ίντα η 11 κατέπεσε γιατί εγκρίθηκε 97 ίντα 11 Κατέπεσε η 11 λοιπόν. Τζούρι 4 και αυτή καταπίπτει. Το δεύτερο τμήμα επίσης. Πάμε στην 99. Βιτάλ Μορέλα, Τζολάινε, Ρομπέρτο Γκουαλτία Ρίπερ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 Ραντζέλ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 Ραντζέλ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 101 ραντζέλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ίντα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ίντα 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε λοιπόν τώρα στη Λίμπε 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική πύλη λατινικό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και πάμε στην ίντα 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ κατά Νομίζω πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Δεκατής ψηφία εναντίον, δέκα υπέρ, μία αποχή. Ψηφίζουμε τροπολογία 110 μπρόκ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 ρανζέλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 ζολάινεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 ζολάινεν υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 3, ζωλά έναν και άλλον Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 ψήφοι κατά 10 υπέρ μία αποχή. Τροπολογία 4 και 5 έχουν καταπέσει. Α, ψηφίζουμε. Τροπολογία 4, Fox υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Σίγουρα εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Λάινεν Μάρτιν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απεσύρθη 11. Πάμε στη 10 ντάφ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 12 φόξ υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τροπολογία 14 Λάινεν Μάρτιν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας σου. Η ισοψηφία δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεν ψήφισατε όλοι φαίνεται όχι ψήφισατε Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 18 υπέρ, 4 ψήφια εναντίον, μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στο συνάδελφο Ραντζέλ για την μακρά καρποφόρα θετικά, θετική εργασία του. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Γκουρμάη. έκθεση Γκούρμαη. Ε, κύριε Χέφνερ, θέλετε να πάρετε το λόγο για την έκθεση Γκουρμάη. Ορίστε. Thank you, Chair. Ε, Όπως είπα χτες, θέλω να κάνω μια προφορική τροπολογία, πολύ σύντομη, για τη συμβαστική 8 λέει η ώρα των ερωτήσεων με την Επιτροπή θα γίνει σε κάθε ολομέλεια για 90 λεπτά για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα οριζόντια θέματα. Τι εννοούμε. Μπορεί να προκύψει μια κατάσταση όπου δεν είναι ένα πόνο αλλά δύο τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι η νέα μορφή της ώρας των ερωτήσεων και θα μπορούσαμε να αφήσουμε τη δυνατότητα στη διάσκεψη των πρόεδρων να πει δεν είναι ένα μόνο αλλά δύο θέματα. Να μην αφαιρέσουμε μέσω των κανόνων του εσωτερικού μας κανονισμού αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό κάνω αυτή την προφορική τροπολόγηση. Κανείς. Τι λέει η κυρία Γκουρμάη. Ναι, άκουσα. Δυστυχώς δεν την υποστηρίζω. Όπως σας είπα υπάρχουν τέσσερις ε, προφορικές τροπολογίες και ελπίζω να με στηρίξετε για αυτές. Να διευκρινίσω, λέει ο κύριος Χέφνερ, η προφορική μου τροπολογία που έστειλα χθε ήταν να υπάρχει πληθυντικό, εδώ, όχι ενικό θέματα, όχι θέμα, αλλά με βάση την απάντησή σας προτείνω να μην αποφασίσουμε αν θα είναι ενικός ή πληθυντικός, να αφήσουμε τον ενικό αλλά να επιτρέψουμε και τον πληθυντικό. Γι' αυτό η προφορική μου ε, τροπολόγηση είναι τώρα ένα ή περισσότερα. Αλλά αν εντάξει το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, εντάξει. Να καταλάβω ποια είναι η θέση της εισηγήτριας, η αντίρρησή της αφορά την πρόταση τροπολογίας που, ψηφ... που θα ψηφίσουμε ή έχετε επί της ουσίας αντίρρηση. Πρέπει να διευκρινίσετε τη θέση σα αυτό δεν έχω καταλάβει. Ποια είναι η θέση τη εισηγήτρια ακριβώ. Σε τι ε, συνίσταται η αντίρρησή της. Δεν είμαι και πολύ υπέρ τη προφορική τροπολογία, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί, να δώσει την εντύπωση ότι είναι υποχρεωτικό να έχουμε πολλά θέματα σε κάθε περίοδο ερωτήσεων προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό είπα όχι. Βέβαια, αν το αναδιατυπώσουμε και πούμε ένα ή περισσότερα θέματα, εντάξει αλλά όταν λέμε ειδικά οριζόντια θέματα, δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα φάσμα διαφορετικών θεμάτων που θα πρέπει να συζητηθούν στην ίδια περίοδο ερωτήσεων. Αλλά εντάξει, αν βάζετε και ένα ή περισσότερα, συμφωνώ. Δηλαδή ουσιαστικά ψηφίζουμε και το βάζουμε στην συμβαστική α, έτσι. Έτσι γίνεται δεκτή. Συμβιβαστική α λοιπόν, αυτή ψηφίζουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που μα λέει η Γραμματεία, θα ψηφίσουμε πρώτα αν θα συμπεριλάβουμε την τροπολογία Hefner στη συμβαστική και μετά θα ψηφίσουμε τη συμβαστική. Έτσι συμφωνείτε, εκτό αν κατάλαβα λάθο. Ποιο είναι υπέρ συμπερίληψη προφορική τροπολογία συμβαστική Α. Σηκώστε το χέρι, παρακαλώ. Κατά. Καλώς. Καλά κατάλαβα λοιπόν. Ψηφίζουμε τη συμβιβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε μπορούμε να πάμε στην τροπολογία 8. Συμβαστική, ε, τροπολογία 8. ΔΑΦ. Μου έφεραν λοιπόν τον τελευταίο κατάλογο που ήρθε χθε το βράδυ. Πάμε ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία Γκούρμα όσον αφορά το άρθρο 116. Ποιο είναι υπέρ. Σηκώστε το χέρι. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Ντάφ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Ενίσταμε εντόνως και αφαιρεί το Συμβούλιο από τους αποδέκτες των από τη θέση του αποδέκτη των ερωτήσεων. Και αυτό δεν το συζητήσαμε καν στην Επιτροπή. Αυτό λέει, αυτό λέει ουσιαστικά αυτή η τροπολογία. Αποκλείει το Συμβούλιο από τον κατάλογο των συνομιλητών μας ουσιαστικά. των ατόμων προς τους οποίους αποτείνουν τις ερωτήσεις μας. Κάτι που είναι τελείως παράλογο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πολιτικό σκεπτικό πίσω από αυτήν την τροπολογία, αλλά δεν το συζητήσαμε. Επίσημα λοιπόν ενίσταμε στην υποβολή αυτής της τροπολογίας. Η κυρία Γκουρμάη. Καλά, να δικαιολογήσω την τροπολογία μου. Ο χρόνο ερωτήσεων προς το Συμβούλιο δεν προβλέπεται στι συνθήκε και μέχρι στιγμής δεν έχει ουδέποτε εφαρμοστεί. Θα προτιμούσα λοιπόν να το αφαιρέσουμε αυτό το σημείο γιατί θεωρώ ότι οι διαδικαστικοί κανόνε δεν είναι η κατάλληλη μέθοδο για να περιλάβουμε ένα τέτοιο πολιτικό μήνυμα ή να επιβάλλουμε υποχρέωση σε άλλο θεσμικό όργανο. Γι' αυτό κατέθεσα τη σχετική προφορική τροπολογία. Ελπίζω τελικά να με υποστηρίξετε. Chairman. Chairman, an oral amendment. Μια προφορική τροπολογία μπορεί να κατατεθεί μόνο όταν υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των μερών. που έστω και ένας ενίσταται, τελεία και παύλα. Πρέπει να προχωρήσουμε. Χρειάζονται δύο μέλη. Ποιος υποστηρίζει την πρόταση ΤΑΦ. Όχι, πρέπει να είναι ομόφωνη αποδοχή μια προφορική τροπολογία. Αν επιμένετε όμω, εντάξει, εγώ υποστηρίζω τον Άντριου Νταφ. Καλώ, αν έτσι έχουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Γκουρμάι. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 8. Νταφ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 ταφ Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 γκουρμάι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, προφορική τροπολογία γκουρμάι. Που αφορά το άρθρο 117. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 μισό λεπτό καταπίπτει 11 και η 12 τροπολογία 12 γκουρμά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 γκουρμάι υπέρ Πρέπει να ψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 15 είναι αυτή που καταπίπτει. 14 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. 18 δαφ υπέρ. Κατά. Πρέπει να κάνουμε επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Να δούμε τα αποτελέσματα. Εγκρίνεται 12 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι εναντίον, μία αποχή. 19 γκουρμάι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 γκουρμάι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Μου λένε ότι ψηφίστηκε συμβαστική Β. Συμπεριλαμβάνεται. Τι ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αποσύρθηκε 32, 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 γκουρμάι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 35. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 κατά πίπτη, 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φτάνουμε στο τέλος αυτής της ψηφοφορίας προφορική τροπολογία της κυρίας Γκουρμάη που αφορά την παράγραφα 2 της αποφάσεως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και άλλη προφορική τροπολογία που αφορά την παράγραφο 3 της αποφάσεως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική για την έκθεση άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Νομίζω ναι. Όποιος θέλει ψηφίζει. Λοιπόν, 18 υπέρ, μία ψήφος εναντίον, μία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην κυρία Γκουρμάη. Μας μένει η έκθεση Σόλτς. Ο κύριος Μπροκ, έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε που δεν το είπα προηγουμένως, αλλά έχω την εντύπωση ότι η ζωή των βουλευτών είναι όσο πιο περίπλοκη. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτή την έκθεση γίνονται ακόμη πιο αδύνατα τα δικαιώματα των βουλευτών, γι' αυτό την καταψήφισα, αλλά ε, είμαι μόνο μία ψήφος. Σας ευχαριστώ. Σημειώνουμε την παρατήρησή σας. ο πρόεδρος. Μπορούμε να προχωρήσουμε να διεξαχθεί η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη συμβαστική ε. Υπέρ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Κατά. αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρα, Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι 13 ψήφοι κατά, 10 ψήφοι υπέρ, μία αποχή, άρα δεν εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε συνεπώς την τροπολογία 11 Σόλτς. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Υπέρ. Κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε ήσυχοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-10. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Επαναλαμβάνει την ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται για μία ψήφο 12-11 και μία αποχή. Η συμβαστική λοιπόν G δεν εγκρίνεται, άρα πρέπει να ψηφίσουμε τη συμβαστική Y Υπέρ, σηκώστε το χέρι παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα καταπίπτουν η, τροπολογία 12-13. Ψηφίζουμε την τροπολογία 12, Ραντζέλ. Υπάρχει προφορική τροπολογία να θέσω. Για τη 12 λοιπόν. Η τροπολογία 12 λέει ο Ραντζέλ θεωρεί ότι η Τρόικα μπορεί να θεωρηθεί ως μία λύση ανάγκης ε, και τελευταία καταφυγή για να, για να λυθεί το πρόβλημα της Ευρωζώνης, αλλά από τούδε και ως το πρέπει και τα λοιπά, αλλά επαναλαμβάνω. Το αρχικό κείμενο της τροπολογίας λέει, θεωρεί ότι η Τρόικα αιτιολογεί το ως μία αναπληρωματική και λύση ανάγκης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της Ευρωζώνης και να λυθεί το πρόβλημα της οικονομικής ε, και χρηματοδοτικής αλληλεγγύης, αλλά και τα λοιπά συνεχίζει. Εγώ θα πρότεινα, θεωρεί ότι, ότι η Τρόικα δημιουργήθηκε ως μια εναλλακτική λύση και λύση ανάγκης και το υπόλοιπο ε, ως έχει αντί να λέει ότι αιτιολογεί το ως εναλλακτική, να λέει ότι δημιουργήθηκε, όχι ότι αιτιολογείται για να λυθεί η προσπάθεια της Ευρωζώνης. Είναι ουδέτερη διατύπωση. Για, με αυτόν τον τρόπο θα υπήρχε ευρύτερη στήριξη αυτή την τροπολογία χωρίς να αλλάζει την ουσία ε, αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Είναι εκτός μικροφώνου δυστυχώς ο πρόεδρος και δεν τον ακούνε οι διερμηνείς. Ψηφίζουμε με τη συμπερίληψη της προφορικής τροπολογίας την τροπολογία 12 Ραντζέλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 Δεν ψηφίζουμε τη 13, διότι καλύπτεται από την συμβαστική Ι, συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, κατέπεσε η 14, πάμε στη 15, ρανζέλ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. così all'emendamento. Πάμε στην τροπολογία 16. Ψηφίζουμε την τροπολογία 16 υπέρ. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 είπε κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να κάνουμε έλεγχο επαλήθευση λοιπόν ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας αποτέλεσμα είναι απόρριψη για μία ψήφο Ανθρωπολογία 18 Ρανζέλ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν λοιπόν οι 20 και 21. Και πάμε στην τροπολογία 22. Ε, μάλλον στην 23 Σόλτς υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω αν θέλετε κάνουμε επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την τροπολογία 23 Σόλτς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτοτε με 13 ψήφους κατά και 10 υπέρ. Συμβαστική κάπα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, καταπίπτει 24, ψηφίζουμε την 25 σόλτς υπέρ, κατά, αποχές, αν θέλετε κάνουμε επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση, ξεκινάει. Ψήφισατε όλοι. Πέρας απορρίπτεται για μία ψήφο. Τροπολογία 26 Σόλτσιπερ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ξεκινάει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι, όχι ακόμα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται για μια ψήφο διαφορά. Τροπολογία 28 Σόλτσιπερ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΙΤΑ. Υπέρ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη συμβιβαστική ΙΤΑ. Ξεκινάει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 14 ψήφοι εναντίον, 9 υπέρ. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται, έτσι νομίζω. 31 υπέρ. Όχι. Ε, Άρα πάμε στην 32 Σόλτσιπερ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 32 Σόλτς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται μία ψήφος διαφορά. Favorevoli. 34. Για την 34. Υπέρ. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Trentasei ancora. Favore. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει 37, οπότε πάμε στην 1, Σόλτσιπερ. Κατά, αποχές εγκρίνεται 2 Σόλτσιπερ. Κατά, αποχές εγκρίνεται 3 Σόλτσιπερ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει συνεπώς η 4. Συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την 5 όμως υπέρ κατά, μάλλον απορρίπτεται. Κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση όμω. Ξεκινάει για τροπολογία 5 Σόλτς. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ. Λοιπόν, συμβαστική C ψηφίζουμε. Κατά. Απορρίπτεται, σίγουρα. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 ρανζέλ υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 7 καταπίπτει, τροπολογία 9, αφορά μόνο τα κράτη-μέλη, είναι προσθήκη στη συμβαστική C υπέρ, κατά, άποχες, νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ξεκάθαρα. Η τροπολογία 9. Η 10 τώρα. Ψηφίσουμε τη 10. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Σίγουρα. Θέλετε να κάνουμε επαλήθευση. Ηλεκτρονικός έλεγχος, η τροπολογία 10 Σόλτς. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Τροπολογία 10, έτσι, τελευταία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 αντίον 9 επέρ μια αποχή. Τελική ψηφοφορία και αυτή με τον ηλεκτρονικό τρόπο που ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Πέρασε το κείμενο. Ε, ευχαριστούμε λοιπόν και συγχαίρουμε τον συνάδελφο Σόλτς. Η ώρα των ψηφοφοριών λοιπόν πέρασε, τις ψηφοφορίες στην ώρα μας και μπορούμε να πάμε στην κανονική συνεδρίαση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

Allora, intanto sul Όσον αφορά το σημείο 15 που αφορά ανακοινώσει αφορά τα αποτελέσματα τη συντομότητα της συνεδρίας των συντονιστών, είναι πολύ σύντομο αυτό που έχω να πω, διότι ουσιαστικά πήραμε αποφάσει μόνο επί δύο σημείων. Το ένα αφορά την προβλεπόμενη ακρόαση για το μέλλον της Ευρώπης 17 και 18 του Μαρτίου αποφασίσαμε κατά κάποιο τρόπο ότι μεταμορφώσουμε. Μπορούμε να συναντήσουμε την επισκεπτή. Ο Βρετανός Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων θα επισκεπτόταν την Επιτροπή μας, αλλά δεν θα ήταν σωστό να ακούσουμε μαζί με άλλους πανεπιστημιακούς και λοιπά και τον Υπουργό και εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. Θα ακούσουμε ξεχωριστά λοιπόν μία μέρα τον Υπουργό θα δούμε, θα μας πει εκείνο το 17 ή 18, ο αρμόδιος υπουργός για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και για το μέλλον της Ευρώπης, ξεχωριστά ο καθηγητής Βάιλερ που είναι πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Ευρωπαϊκού που δέχτηκε, θα μιλήσει και κάποιος θα αναφερθεί στο νέο σύμφωνο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και μας έστειλε ένα έγγραφο είναι το Ίδρυμα ε, Μπελταζίνο μαζί με έναν άλλο φορέα και μας έστειλαν ένα έγγραφο, Είστε ένα έγγραφο στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου που αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Θα τους ακούσουμε λοιπόν αυτούς και θα ακούσουμε τι έχουν να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Δεύτερον, το θέμα της Ευρωπα... η της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των μυρωδών δικαιωμάτων. Από την αρχή της θητείας έχουμε εργαστεί επί του θέματος σαν Επιτροπή, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου της Ευρώπης. Θέλουμε να γνωρίζουμε περισσότερα και θα υποβάλουμε μία ερώτηση ούτω ώστε να έχουμε επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το θέμα αυτό. Εάν το δέχεστε, θεωρείται ότι είναι η λιμένη απόφαση. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο, πριν τα διάφορα, που είναι η τροποποίηση του κανονισμού του Κοινοβουλίου, που προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ε, με μπερδεύουν λίγο οι ημερομηνίε. Ε, η συνάντηση με τον Υπουργό είναι 17 Μαρτίου. Και μετά τι είπατε? Μια συνάντηση με τον καθηγητή ποιον? Βάιλαντ. Βάιλερ. Α, πότε. Α, την επόμενη 18. Ναι, έτσι αποφασίστηκε, ναι. Δε, θέλουμε να είναι ξεχωριστές αυτές οι δύο συναντήσεις, να αποφύγουμε συγχύσεις. Αν είναι διαθέσιμος ο κύριος Υπουργός να έρθει στις 17, θα τον ακούσουμε στις 17, αν είναι διαθέσιμος στις 18, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και να κάνουμε στις 17 τη συνάντηση με τον καθηγητή Βάιλερ και τους άλλους ε, πανεπιστημιακούς. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Πρέπει να είναι όμως ξεχωριστές εκδηλώσεις όσον αφορά την, το πότε θα μπουν, πότε θα, θα, θα ξεκαθαρίσουν το θέμα του πότε θα διεξαχθούν οι ακροάσεις. Τόσον αφορά τον κανονισμό για την να επιτραπεί η ηλεκτρονική υπογραφή στο Κοινοβούλιο, εκεί διορίστηκε η συγητή ο συνάδελφος Σέπφλιν, τον οποίον καλό να πάρει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια τεχνική τροπολογία που ουσιαστικά επιτρέπει την διανομή εγγράφων, είναι πιλωτικό πρόγραμμα, καθώς και το θέμα των ηλεκτρονικών υπογραφών αρκεί να έχει εξασφαλιστεί τεχνική αξιοπιστία και ορθότητα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να βάζουμε ηλεκτρονικές ε, υπογραφές ε, στα έγγραφα. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο? Αν είναι τόσο απλό και τόσο σαφές μπορούμε να θέσουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες 27 Φεβρουαρίου, προθεσμία υποβολή τροπολογιών μέχρι το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί το θέμα στην ε, συνεδρίαση στις 18 Μαρτίου. 18 Μαρτίου η ψηφοφορία. Ούτως αποφασίσαμε και στα διάφορα δεν έχω τίποτα. Ε, δεν βλέπω να έχει σηκωθεί χέρι. Σας πληροφορώ ότι λέω Δευτέρα 17 από τις 15 μέχρι 18 και 30 θα είναι η επόμενη συνεδρίαση και την επόμενη μέρα θα συνεχιστεί από 9 μέχρι 12 και 30 στις 18 Μαρτίου, 17 Μαρτίου το απόγευμα 18 Μαρτίου το πρωί. Ευχαριστώ όλους. Πέρασε η συνεδριά σας. Σας ευχαριστούμε και γεια σας. squadra negoziale stasera? Sì, sì, eh, sì, sì stasera alle, alle 5 credo. Ricordo, scusate, e la vicepresidente Gourmai mi ricordo una cosa. Μου υπενθυμίζει κάτι σημαντικό το κυρία Γκουρμάη. Φτάνουμε... Φτάνουμε στο τέλος της εκθέσεως όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων των Πολιτικών Κομμάτων. Και αύριο θα πρέπει να διεξαχθεί ο τριμερής διάλογος θα πρέπει να συναντηθούμε την πραγματευτική ομάδα στις 4 θα συναντηθούμε. Με εκείνους που συμμετέχουν στην πραγματευτική ομάδα παρακαλούμε λοιπόν αυτοί που είναι στην ομάδα να είναι στην αίθουσα «5Ε2» ε στην αίθουσα 5Ε2 ε στις 4. Ευχαριστώ. Πέρα συνεδριά σου στο επανειδή.